Δικαίωμα στο νερό. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ήταν το πρώτο παράδειγμα επιτυχούς δημοκρατικής προσπάθειας και χρειάζονταν 1,8 εκατομμύρια υπογραφές, αλλά συνελέγησαν τελικά και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης είναι βασικό δικαίωμα για τους πολίτες και δεν μπορούμε να ε, το παραγνωρίσουμε. Στην Ιρλανδία, όπως ξέρετε, έχουμε τέλη που μας έχουν οδηγήσει στις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες που γνώρισε ποτέ η Ιρλανδία για αυτό το ζήτημα και ε, θεωρούσαμε ε, τότε ότι ήταν ένας ε, ένα προοδευτικό τέλος, έτσι θεωρούσε η κυβέρνηση. Κατα, καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση των πολιτών. Παρά την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών άνευ προηγουμένου, η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ανεπαρκής και δεν ανταποκρινόταν ε, στις ε, ανάγκες που είχαν προκύψει από την καμπάνια που έκαναν οι ίδιοι οι πολίτες. Μέσα στην έκθεση προσπάθησα να δώσω μια πιο ικανοποιητική απάντηση στους πολίτες. Περιμένουν ε, μια προσφορότερη δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχει κατατεθεί καμία νομοθετική πρόταση που καταχειρώνται σαν οικονομικό δικαίωμα το νεροίδρευση και αποχέτευση για τους πολίτες. Αυτό το δικαιούνται οι πολίτες μέσω από αυτής της πρωτοβουλίας και του έχει αγνοήσει προ το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ μέσα από την έκθεσή μου λοιπόν να διορθωθεί αυτό το λάθο ε, και ε, ο ανταγωνισμό ανάμεσα στι ιδιωτικέ επιχειρήσει ε, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στο παρελθόν και ούτε και πρόκειται σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό το νερό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι και κερδοσκοπικές αυτές οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται το νερό και ε, είναι κέρια σημασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει τα δικαιώματα των κρατών μελών να οργανώνουν όπως ε, κρίνουν προσφορότερα τις υπηρεσίες τους, ε, υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης. θέλουμε όταν αρχίσουν να διαχειρίζονται και πάλι αυτές τις υπηρεσίες και μην ξεχνάμε ότι μετά την πανταγώδη επιτυχία ιδιωτικών επιχειρήσεων σε αυτό το τομέα τελικά επανεθνικοποιήθηκαν αυτές οι υπηρεσίες σε πολλές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την υποστήριξη των βουλευτών από τις πιο προοδρευτικές ομάδες. Έχουμε την υποστήριξη και με απογοητεύει ε, το ΕΛΚ. Μην ξεχνάμε ότι και οι συντηρητικοί έχουν ένα εναλλακτικό ψήφισμα όπου τονίζουν τα κύρια σημεία της έκθεσής μου και βλέπω ότι ε, προσπάθησαν ε, να κρύψουν αυτήν την ντροπή, αυτή την επέσχυντη στάση τους. Προσπαθούν να αποδυναμώσουν τις τροπολογίες της, ε, την έκθεσή μου και ε, ε, προσπαθούν να καταργήσουν την κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν έχει αναλάβει καμία δράση, επειδή δεν έχει κατοχυρώσει ως οικονομικό δικαίωμα το δικαίωμα στο νερό και δεν μίλησαν καθόλου για τα κρατικά μονοπόλια και θέλουν να παραμείνουμε ουδέτεροι ως προς την ανάγκη απαγόρευσης της ιδιωτικοποίησης σε αυτού του τομέα Επίσης, ε, διαγράφουν την αναφορά ε, στην ε, στην ΤΙΤΗ, διότι θέλουμε να εξαιρεθούν ρητά αυτές οι υπηρεσίες ε, από αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, και οι συντηρητικοί ε, φυσικά υποστηρίζουν το ΕΛΚΑ. Είναι πραγματικά ντροπή, διότι 2,1 εκατομμύρια πολίτες ζήτησαν να κατοχυρωθεί αυτό το βασικό τους δικαίωμα. Είναι η μοναδική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί σε αυτήν τόσο επιτυχημένη πρωτοβουλία των πολιτών. Καταλαβαίνετε πόσο θα καταστρέψει αυτό την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν τελικά εγκριθεί αυτό το εναλλακτικό συντηρητικό ψήφισμα που δεν υποστηρίζεται από την καμπάνια που έκαναν οι ίδιοι οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμη να σταθεί στο πλευρό των πολιτών. Εάν περάσει αυτό το ψήφισμα θα πνιγούν οι συντηρητικοί ε, στο ίδιο τους το ψήφισμα. Σας ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριος Τζάκοβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προέρχομαι από μια μικρή περιφέρεια στη Δυτική Κροατία και θα μπορούσα να σας δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες ίδρευσης που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των πολιτών. Το νερό αποτελεί έναν απόσπαστο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ένα 99% των ανθρώπων στην περιφέρειά μου έχουν ε, πρόσβαση σε υπηρεσίες ίδρυυσης μέσω μιας δημόσιας εταιρείας ίδρυυσης. Έχουμε επίσης ε, εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και μια πολιτική αλληλεγγύης απέναντι στους πολίτες. Ανήκω στην ομάδα των φιλελευθέρων, αλλά είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης ε, των υπηρεσιών υδροδότησης. Πιστεύω ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νερό και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά αντιτίθεμαι εδώ πέρα στη γενικότερη τάση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι μπορούμε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό όταν αυτό διατίθεται μόνο μέσω μιας δημόσιας υπηρεσίας. Ο κύριος Τούρμες για ένα λεπτό. Ε, Εκατομμύρια πολίτες έχουν προσυπογράψει αυτό για το νερό το δημόσιο αγαθό που δεν πρέπει να φιλελευθερωποιηθεί, απελευθερωθεί, δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανταγωνισμού ή κερδοφορίας και πρέπει να μπορέσουμε να αποφύγουμε επιχειρήσεις να εμπλακούν στην εκμετάλλευση του νερού, του υδάτινου αυτού πόρου σκεφτόμουν ότι υπάρχει πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο για να υποστηριχθεί αυτό το αίτημα όπως συμβαίνει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θλίβομαι ιδιαίτερα για αυτό το οποίο συνέβη με τους συντηρητικούς και το ΕΛΚΑ και το ECR που θέλουν οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την εκμετάλλευση του νερού και να ζητήσουν να απελευθερωθεί η χρήση, η εκμετάλλευση του νερού και στην Ευρώπη και στην TTIP, στην Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων ε, όσον αφορά τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γίνεται λόγος για την μη ιδιωτικοποίηση του νερού Προέδρου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της που περιλαμβάνει όλα όσα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στην ημερίδα που διοργάνωσε το κίνημα «Σώστε το νερό» στη Θεσσαλονίκη τον προηγούμενο Μάιο που είχαμε εκληθεί ως ομιλητές. Στηρίζω και εγώ με τη σειρά μου τον αγώνα των κινημάτων και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών για το δικαίωμα στο νερό και εφιστώ την προσοχή στην Επιτροπή να εξαιρέσει τις υπηρεσίες ίδρυυσης από τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ttip και την tisa και η ευρωπαϊκή ένωση να τηρήσει τη συνθήκη και να μην προωθεί την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ίδρυυσης ιδίως σε χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο όπως συμβαίνει στην ελλάδα με την ειάθ στη θεσσαλονίκη. στηρίζω την έκθεση και αντιτάσσομαι στις τροπολογίες του ελκ που προσπαθεί να αποδυναμώσει την έκθεση και την καμπάνια των ευρωπαίων πολιτών. το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό και η πρόσβαση στην ίδρυυση και την αποχέτευση αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη όπως καθορίζει και η ίδια η γενική συνέλευση του οηε. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπόιλαν για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση. Προέρχομαι από την Ιταλία όπου οι 27 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν σε δημοψήφισμα προκειμένου το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Αλλά δυστυχώς το δημοψήφισμα αυτό δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, δικαίωμα στο νερό, να μην αντιμετωπίσει την ίδια κατάληξη. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, δικαίωμα στο νερό. Και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει προ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει αυτό που τα ίδια τα Έθνη έχουν αναγνωρίσει ως αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα, η πρόσβαση στο νερό. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα αυτό ως αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Για λόγους δημοκρατίας, για λόγους λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πραγματικά να τηρήσει το περιεχόμενο αυτής τη Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ελπίζω να καταφέρει να συμβάλλει και η ε, ομάδα που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαρνό για ένα λεπτό παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ. Τι να πω, δεν ξέρω πώς να ψηφίσω, διότι συμφωνώ με ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που μας λέει η συγγήτρια. Συμφωνώ, είναι ανθρώπινο δικαίωμα το νερό. Συμφωνώ ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από την διατλαντική ε, ε, συμφωνία TTIP. Δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμο αυτό φυσικά, πρέπει να είναι κρατικό μονοπόλιο το νερό. Αυτό πιστεύω προσωπικά. Και συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίε που έχει η συγγήτρια για την βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες για το νερό. Έχουμε και 1,2 εκατομμύρια υπογραφές ε, για αυτή την πρωτοβουλία και παρόλα αυτά ε, δεν γίνεται η συζήτηση που θα έπρεπε. Εγώ συμφωνώ με τη στήριξη των ΟΤΑ και το, για το ρόλο τους για τη διαχείριση του νερού. Όμως ε, θα πρέπει να αποφασίζω και πώς θα, πληρώ, πώς θα ψηφίσω γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να ζητώ, ε, ζητούμε χρηματοδότηση. Εγώ θα σας έλεγα να περιμένετε να κοιμηθείτε και θα σας έρθει η ιδέα πώς να ψηφίσετε αύριο το πρωί. Ας ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο για να απαντήσει. Ευχαριστούμε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ε, εύχομαι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα την κυρία Μπόιλαν για τη συνέχεια που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Δικαίωμα στο Νερό. Όπως κατέστησε σαφές στην απάντηση σε αυτή την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νερό δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν όπως άλλα προϊόντα, αλλά μια κληρονομιά που πρέπει, ένα αγαθό που πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί η πρόσβαση στο νερό ως δεδομένο δικαίωμα παρότι πολλοί το κάνουν αυτό στην Ευρώπη. Πάντα τόνιζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια σημαντική προϋπόθεση για την ελεύθερη πρόσβαση στο νερό είναι η διασφάλιση και προστασία των υδάτινων πόρων. Είναι αυτό ακρογωνιός λήθος της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος. Η οδηγία για το πόσιμο νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η αντιμετώπιση των απόνερων και της, ε, την υγειονομική βάση που αποτελεί τη βάση για την ενσωματωμένη αντιμετώπιση, ολοκληρωμένη ε, αντιμετώπιση του νερού. Πρόσβαση στο νερό και η ε, υγειονομική διάσταση έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Με την διακήρυξη της χιλιετίας με τα στατιστικά στοιχεία δείχνει ότι πάμπολοι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες υγειονομικές ε, υποδομές και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το στόχο της ε, διαθεσιμότητας και της αηφορίας στη διαχείριση του νερού προς όφελος όλων βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας στο θεματολόγιο της ε, στρατηγικής μετά το 2015 και θα πρέπει να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στις εξωτερικές μας δράσεις και στις εσωτερικές μας πολιτικές και δράσεις για το νερό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αναγκαία εκείνη όθηση ώστε με τους εταίρους μας να μπορέσουμε στο ε, άμεσο μέλλον να σημειώσουμε πρόοδο. Θέλω να τονίσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στη διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και τα υγειονομικά ως υποδομές. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του νερού ως δημόσιου αγαθού. Η διαθεσιμότητα και οι υπηρεσίες ε, όσον αφορά το νερό αποτελούν ευθύνη των τοπικών αρχών, μια και βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσαφηνίσει την αρχή της ουδετερότητας. Οι κανόνες των συνθήκων απαιτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αμερόληπτη όσον αφορά τις ε, κρατικές αποθε... Ε, αποφάσεις, όσον αφορά την... το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το νερό επίσης ε, οι άδειες που θα χορηγούνται θα αναγνωρίζουν ε, τον ιδιαίτερο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού, ιδιαίτερα για το πόσιμο νερό και τα υγειονομικά που έχουν αποκλειστεί όσον αφορά τα αγαθά υποεκμετάλλευση, καθώς επίσης ε, και την επιλογή των μεθόδων διαχείρισης του νερού που έχει αναγνωριστεί ως αρχή κανέ, καμιά εμπορική συμφωνία δεν έχει περιορίσει τις ελευθερίες να διοργανώνουν τα κράτη-μέλη τις δημόσιες υπηρεσίες τους με το νερό συμπεριλαμβανόμενο ώστε να μπορούν να δρουν ελεύθερα. Και η TTIP, η Διατλαντική ε, Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου δεν θα κάνει τίποτα το διαφορετικό. Επιπλέον επιβεβαιώνω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δράσεις που θα διασφαλίζουν ότι αυτές οι αρχές θα είναι στον πυρήνα, στην καρδιά των πολιτικών και θα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σπουδαιότητα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι πολιτικές αυτές να βελτιώνουν την πρόσβαση στο νερό και στα υγειονομικά ως υποδομές για το σύνολο του πληθυσμού στις περιβαλλοντικές πολιτικές και τη χρηματοδότησή τους. Τώρα θέλω και πάλι να υπογραμμίσω τη θετική επίπτωση που έχει η πρωτοβουλία πολιτών για το δικαίωμα στο νερό θέτοντας ψηλά στο θεματολόγιο, στην ημερήσια διάταξη τις προτεραιότητες αυτές. Καλωσορίζουμε τις προοπτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξετάζει προσεκτικά αυτές τις προοπτικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάληψη πρωτοβουλειών, για την οδηγία για το πόσιμο νερό για παράδειγμα για την ε, αναθεώρηση του πλαισίου για το νερό και τον διάλογο που εξελίσσεται, βρίσκεται υπό εξέλιξη με τους εμπλεκόμενους και την κοινωνία των πολιτών για τις βέλτιστες προοπτικές για το νερό και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται. Ολοκληρώνοντας, θέλω να προσθέσω ένα σημαντικό στοιχείο. Οι πολιτικές για το νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το παρελθόν ε, δημιούργησαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν δυνατότητες παροχής του νερού με τις αναγκαίες υποδομές τους πολίτες. Παραμένουν όμως οι προκλήσεις. Πρέπει να δράσουμε νομοθετικά αλλά και με στοχοθετημένες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα προετοιμάσουμε. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις διατάξεις και ρυθμίσεις για το νερό πανευρωπαϊκά. Επίσης ε, η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καλοδεχούμενη ιδιαίτερα για αυτές τις δράσεις και την εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών για ε, χάρη στη μεγαλύτερη διαφάνεια που μπορούμε να επιτύχουμε. Η πρόσβαση στο νερό και η υγειονομική συνιστόσα είναι πολύ σημαντικές διαστάσεις και θα ληφθούν υπόψη στο, το μελλοντικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία βρίσκεται εδώ και μια καινούρια, μια καινοτομία που εισήχθη με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εμπλέκονται και συμμετέχουν έτσι οι πολίτες στην ανάπτυξη του θεματολογίου και των δράσεών μας. Υπάρχει όμως ακόμα περιθώριο για βελτιώσεις. Στην έκθεση για την εφαρμογή 211 κάθετος 2011 για την πρωτοβουλία των πολιτών όσον αφορά τη δημοσίευση του Μαρτίου 2015 αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τρία χρόνια εφαρμογής του τι είχε συμβεί ταυτοποίησε αρκετά θέματα η έκθεση αυτή ως θέματα που πρέπει να αποτελέσουν βάση περαιτέρω συζήτησης και προβληματισμού για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Αναμένει τώρα προτάσεις από τους εμπλεκόμενους και όσους συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις ε, δράσεις. Αυτή η έκθεση θα ενταχθεί στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δράσεις και η λειτουργία της πρωτοβουλίας των πολιτών να γίνει αυτή η πρωτοβουλία το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δοθεί συνέχεια λοιπόν έτσι στην μετεξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο την έκθεση αυτή συνάδελφοι. Θα πάλι 9 το πρωί.